αλλιώ πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία. Μπορεί να βρείτε αυτέ τι συστάσει στην ιστοσελίδα τη Ολομελία. Και τώρα, πάμε στη διάταξη των εργασιών. Έχουμε το οριστικό. Ε, ε ε, στην ουσιαστική ε, ημερησία διάταξη και σας έχει διανεμηθεί το σχέδιο αυτής όπως αποφασίστηκε από το Προεδρείο και έχουμε επίση και κάποιες ε, προτάσεις τροποποίησης της ημερησίας διατάξεως για την Τετάρτη έχει ζητηθεί ε, να γίνει η ψηφοφορία τη εκθέσεω Κορά όσον αφορά την αυτοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων για την καταχώρηση σχημάτων στην Πορτογαλία. Και αυτό επομένω να ψηφιστεί την Τετάρτη. Αν δεν υπάρχουν ενστάσει, εγκρίνεται η πρόταση τροποποίησεω. Η πολιτική ομάδα, η ΕΝΕΦ, έχει ζητήσει την 5η 8 Φεβρουαρίου ή 5η 1η Μαρτίου να ε, γίνει η ψήφιση Τη εκθέσεως Χιούμπνερ και Περέρα όσον αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να παραστούν στην κηδεία του συναδέλφου Φεράν. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Νίκολας Μπέι για να διατυπώσει το αίτημα αυτό του ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας ε, προς τιμήν του Εντουάρ Φερόν, του εκλειπώντος ε, συναδέλφου μας. Θα ενημερώσουμε την οικογένειά του για αυτά σας τα λόγια. Και ευχαριστούμε πολύ που τηρήσαμε και ένα λεπτό σιωπής. Θα θέλαμε να τροποποιήσουμε την μεσαία διάταξη της Ολομέλειας έτσι ώστε η, η ψηφοφορία της Τετάρτης ε, ε, Σίλβα Περέιρα για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις ευρωεκλογέ και το Brexit, αυτή η ψηφοφορία να γίνεται την Πέμπτη αυτή τη βδομάδα ή στις Βρυξέλλες την 1η Μαρτίου. Ε, επικρατεί διχασμός απόψεων στο Κοινοβούλιο και η απουσία πολλών βουλευτών της ίδιας πολιτικής ομάδας λόγω της ε, κηδείας ε, που θα γίνει στο Παρίσι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε να ε, μετακινηθεί, να αναβληθεί η ψηφοφορία αυτή. Και αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσάρνεσκι, ε, να πω ότι προφανώς ε, δεν συμμεριζόμαστε αυτά που είπε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά υπόθηκαν στο πλαίσιο ενός έντονου διαλόγου με έναν συνάδελφό του και δεν είναι δυνατόν να είμαστε και εμπλεκόμενοι και δικαστές ταυτόχρονα, ε, οπότε νομίζω ότι τα δικαιώματά του έχουν ε, προσβληθεί και παραβιαστεί. Πρόεδρος. Η ε, δημοκρατία, στη δημοκρατία γίνονται σεβαστέ οι αποφάσει πλειοψηφία και η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία. Άλλωστε και η τελική ψηφοφορία θα γίνει από την Ολομέλεια μυστικά και ο καθένα θα αποφασίσει τι επιθυμεί. Θέλει κάποιος τον λόγο κατά του αιτήματο του κύριου Μπέ. Έχετε το λόγο. We should say that the parliament... Θα ήθελα να πω ότι η θέση του Κοινοβουλίου ήταν απολύτως σαφής όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουμε τη θλίψη μας για τους συναδέλφους και για τον συνάδελφο κύριο Φέχα. Παρ' όλα αυτά τώρα ασχολούμαστε με ένα άλλο θέμα δηλαδή δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις στις οποίες έχουμε καταβάλει μεγάλο έργο και όπου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει μια σαφή θέση και να ακολουθήσει και μια ξεκάθαρη ψηφοφορία. Η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών δεν συμφωνεί να αναβληθεί η ψηφοφορία της Τετάρτης. Πρέπει να γίνει η ψηφοφορία την Τετάρτη και θα ήταν σφάλμα να καθυστερήσουμε αυτή την ψηφοφορία, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει μια ξεκάθαρη θέση από αυτόν, πριν από την συνάντηση των ηγετών που θα ασχοληθεί με το ίδιο θέμα. Μας λυπεί ε, το γεγονός του θανάτου του συναδέλφου, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να αναβάλουμε την ψηφοφορία για μια τόσο σημαντική έκθεση. Και τώρα θα ψηφίσουμε όσον αφορά την πρόταση τη πολιτική ομάδα Γενέα που έχουν ζητήσει να γίνει αναβολή από την Τετάρτη στην Πέμπτη, στη δεύτερη. Ε, Συγγνώμη, την, λέω την 1η Μαρτίου, 5η Μαρτίου, στη δεύτερη σύνοδο που έχουμε όσον αφορά το να μπορέσουν αντί να ψηφίσουν την έκθεση Χιούμπνερ Περέρα να πάνε στην κυρία του κυρίου Φερόν συνάδελφου. οποίο είναι υπέρ τη ε, προτάσεω του αιτήματο του κυρίου Μπέ κατά αποχές. Δεν θα τροποποιηθεί η μέρη διάταξη. Τώρα έχουμε την έκθεση Φερνάντε που αφορά την ετησία έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καλώ όρισε ο, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κύριο Μάριο Ντράγκη. Και πριν το δώσουμε το λόγο. Παρακαλώ όποιος θέλει να αποχωρήσει να το κάνει συντόμως.